σας και σας ευχαριστώ εκ νέου για την τη αυτή συζήτηση. Ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ κυρία μου για την σύνοψη που κάνατε τη συζητήσεως. Έχουμε λάβει πέντε προτάσεις ψηφισμάτων για την ολοκλήρωση τη συζήτηση του θέματο αυτού, το, το οποίο συζήτησε λίγη τώρα και προχωρώ αμέσω στην εκφώνηση του επομένου θέματος. Δήλωση δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Το λόγο λαμβάνει πάλι η Επίτροπος κυρία Γεώργιεβα. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που από τον αέρα με κατεβάζετε στη γη, στους σιδηροδρόμους. Είναι προνόμιο για μένα να εμφανίζομαι ενώπιον του Κοινοβουλίου και να μπορέσω να το ευχαριστήσω για την υποστήριξη που προσέφερε στις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να προχωρήσει σε σωστή εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους, που είναι δική τους ευθύνη. Η Κομισιόν συμμορφώθηκε με τις υποχρεώσεις της ως θεματοφύλακος των συνθήκων, στέλνοντας αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις σε 22 χώρες μέλη για μη σωστή εφαρμογή του πρώτου, της πρώτης δέσμης. Και δεν πρόκειται να διστάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες οι οποίες ακόμη δεν συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία να προσφύγει εναντίον των χωρών αυτών μελών ενώπιον του δικαστηρίου. Οι ιδιαίτερες λεπτομέρειες των διαδικασιών αυτών είναι θέμα μεταξύ της Επιτροπής και των χωρών μελών. Πάντως οι υπηρεσίες μας ήδη έχουν υποβάλει στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών πλήρη λίστα όλων των διαδικασιών παραβάση σημειώνουμε και διαπιστώνουμε ότι το επίπεδο επενδύσεων στην υποδομή των σιδηροδρόμων παραμένει ανεπαρκές σε πολλές χώρες μέλη. Ωστόσο δεν συμφωνεί η Επιτροπή με την δήλωση που έγινε ότι δεν έχει κάνει επαρκή παρακολούθηση, επαρκές monitoring η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δέσμη προδιαγράφει ότι οι χώρε μέλη οφείλουν να εξασφαλίσουν ισοσκελισμένο προπολογισμό για τι επενδύσει αυτέ σε εύλογο χρονικό διάστημα. Όπου διαπιστώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή η ρύθμιση, αυτή η διάταξη δεν έχει γίνει σεβαστή από τι χώρες μέλη, έχουν αρχίσει διαδικασίε επί παραβάση. Ορισμένες ομάδες συμφερόντων θέλουν να πιέσουν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει με τη σειρά τη τις χώρες μέλη για να αυξήσουν τις επενδύσεις. Ίσως και εμείς να θέλαμε να δούμε κάτι τέτοιο, αλλά δεν υπάρχει νομική βάση για να υποστηρίξουμε αυτή την απέτηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις πολιτική έκκληση προς τις χώρες μέλη, διότι αντιλαμβανόμαστε τη σημασία των επενδύσεων στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών για να υπάρξει μια βιώσιμη σιδηροδρομική ε, διασύνδεση των χωρών μελών. Και τα είδαμε αυτά και πρόσφατα με, τα, με το κλείσιμο των αεροδρομίων λόγω της ε, ηφαιστειακής που δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν οι άνθρωποι και πόσο χρειαζόταν τα τρένα τα οποία ήταν υπερπλήρη. Θα πρέπει να τεθεί και το θέμα της έλλειψης πόρων. Σας βεβαιώνω ότι οι επικείμενες προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα αναφέρονται ακριβώς σε αυτό. Θα διευκρινίζουν τις αρχές για τις, ε, για τις ε, υποδομές και τα σχετικά τέλη που θα πρέπει να εισπράττονται έχει ξεκαθαρίσει την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πάντως στην ανακοίνωσή της του Μαΐου 2006. Αυτοί που διαχειρίζονται τις ε, υποδομές θα πρέπει να είναι ανεξάρτητοι από, αυτούς, από τις εταιρείες, από τις δρομικές εταιρείες ή τις δρομικές holding. Διότι έλεγχος και ανεξαρτησία δεν πάνε μαζί. Και βασισμένη στην ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηριού, εμείς καταλήξαμε σε συγκεκριμένε αρχές, συγκεκριμένα κριτήρια για την αξιολόγηση της ανεξαρτησίας της ε, θηγατρικής η οποία ασχολείται με τις ε, υποδομές από την μητρική εταιρεία. Το ψήφισμα επίσης ζητεί να εφαρμόζεται η αρχή της αμοιβαιότητας. Αυτό βέβαια δεν είναι αρχή την οποία μπορούμε να δεχτούμε γενικά ως εφαρμογή δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Πρέπει να εφαρμόζονται οι υφιστάμενες κοινοτικές οδηγίες για κάθε χώρα μέλος ανεξάρτητα από το τι κάνουν οι άλλες χώρες. Διότι βεβαίως αλλιώς η πιο αργή χώρα μέλος θα επηρεάζει και τον ρυθμό των υπολείπων. Συμφωνώ λοιπόν με το ψήφισμα σε όσα λέει για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης μέτρων και σας διαβεβαιώνουμε και πάλι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη δουλειά της και εξακολουθεί να επιμένει ότι θα την κάνει. Δεν θα πρέπει να παραμείνει μόνη της βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην προσπάθειά της να ανοίξει την πρόσβαση στις αγορές και στην προσπάθεια αναζωογόνησης του σιδηροδρόμου ως βιώσιμου τρόπου μεταφοράς. Υπολογίζουμε, βασιζόμαστε στην δική σας υποστήριξη, ώστε η πολιτική μας των σιδηροδρόμων να γίνει πραγματική επιτυχία και να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και χάρη σε αυτούς να ξεπεράσει την παρούσα οικονομική κρίση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, συγγνώμη. Σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστούμε για τις πληροφορίες που παρέσχατε. Για δύο λεπτά θα έχουν τώρα τον λόγο οι εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων. Και πρώτος ο κύριος Κάρλο Φιντάντσα, του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι συνάδελφοι. Είναι το ότι για την εφαρμογή της πρώτης δέσμης του συνδυοδρομικών μέτρων καθυστέρησαν πολύ τα πράγματα. Το 2001 εγκρίθηκε η νομοθεσία, η μεταφορά προβλεπόταν μέχρι τις 15 Μαρτίου του 2003 και Εν ώψη τη ανασεώρησης τη πρώτη δέσμη των συνδυροδρομικών μέτρων, θα ήθελα να επισημάνω ότι πέραν του θέματο των επενδύσεων που πολύ σωστά επεσήμανε η, Ευρω... η Επίτροπο, υπάρχουν τρία βασικά θέματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την εφαρμογή τη δέσμη των μέτρων. Καταρχά, από τι διάφορε δυσκολίε που ανέκυψαν τα τελευταία χρόνια, προέκυψαν και κάποια θέματα από νομική σκοπιά ε, για την ανεξαρτησία των διαχειριστών των υποδομών. Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιε περαιτέρω διευκρινήσει επί του θέματο, διότι αυτό ήταν ένα από τα προσκόμματα που αντιμετωπίσαμε τα τελευταία χρόνια και φαντάζομαι ότι ε, στη διάρκεια τη αναδιατύπωση τη πρώτη δέσμη θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία νέα βάση. Δεύτερον, Είμαι βέβαιο ότι η απελευθέρωση των αγορών των σιδηροδρόμων θα πρέπει να θεωρείται ικανή και αναγκαία συνθήκη για όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρουμε ότι όλοι στα λόγια είναι υπέρ της ελευθέρωσης των αγορών, αλλά ε, μετά ε, στην εφαρμογή όλα χωλένουν. Θεωρώ ότι αυτό είναι απαραίτητο για να επιτύχουμε το στόχο της βελτίωσης των σιδηροδρόμων και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, παρακινήσει τα κράτη-μέλη να επιτύχουν αυτό το στόχο. Τρίτον, αυτό το απόλυτο μονοπόλιο που υπάρχει εντός κάποιων κρατών μελών ε, δίνει τη δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να το εκμεταλλεύονται. Και επειδή ακριβώς υπάρχει ο στρατηγικός στόχος της απελευθέρωσης των αγορών, εμείς θεωρούμε και μαζί με τον συνάδελφο Γκρός το έχουμε βάλει στο ψήφισμα το οποίο θα ε, ψηφίσουμε αύριο, ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί η αρχή της αμοιβαιότητας, η οποία είναι απαραίτητη αυτή τη στιγμή προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία του ανοίγματο των αγορών. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο κύριος Ελχαντράουι των Σοσιαλιστών έχει το λόγο. Ορίστε, για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, άμα δείτε το μερίδιο των σιδηροδρόμων στις μεταφορές τα τελευταία 20 χρόνια θα καταλάβετε ότι αντιπροσωπεύει περίπου 10% για τα εμπορεύματα. Και αυτό είναι πολύ χαμηλό ποσοστό. Αν θέλουμε κάτι να κάνουμε χρειάζεται ολόκληρη σειρά μέτρων, όχι μόνο προσωρινών πολιτικών μέτρων αλλά και πολύ τεχνικά θέματα συνδυασμού με άλλους τρόπους μεταφορών, βελτίωσης των υποδομών, ε, ενημέρωσής τους, ε, εκμοντερνισμού τους, εξυγχρονισμού τους δηλαδή κτλ. Και βέβαια αυτά όλα αφορούν τελικά την πρόσβαση στην αγορά. Γι' αυτό είναι τόσο σημαντική η δέσμη μέτρων για τους σιδηροδρόμους. Είχε εγκριθεί για πρώτη φορά το 2001 και έπρεπε μέχρι το 2003 να είχε μεταφερθεί στα κράτη-μέλη, αλλά ακόμη και σήμερα δεν το έχουν μεταφέρει όλα τα κράτη-μέλη στην εθνική τους νομοθεσία και αυτό είναι απαράδεκτο. Η Κομισιόν καθυστέρησε πάρα πολύ Τρία θέματα τίθενται εδώ. Πρώτον χρειάζεται ένα ανεξάρτητο σώμα που να διαθέτει τα κατάλληλα, τους κατάλληλους πόρους για να επιβάλλει την απελευθέρωση του τομέα αυτού πραγματική ανεξαρτησία για να υπάρξει όντως ισονομία και τρίτον χρειάζεται, χρειάζεται λέγω η κατάλληλη υποδομή να εξυγχρονιστεί, το έχω ξαναπεί και πριν. Ώστε οι σιδηρόδρομοι να γίνουν ανταγωνιστικοί ως προς τους άλλους τρόπους μεταφορών. Για την απελευθέρωση θα ήθελα να πω ότι πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα το θέμα της σωστής εφαρμογής της πρώτης δέσμης και για τις μεταφορές επιβατών διεθνώς εδώ χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να χορηγήσουμε υψηλό επίπεδο ε, μεταφορών για τους επιβάτες για να είναι αυτές άνετες και αποτελεσματικές. Πρέπει να είναι αυτό προτεραιότητα και όχι μόνο ένα μέσον μέσα στα γενικότερα πλαίσια της απελευθέρωσης. Σας ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Δύο λεπτά τώρα. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, κατεβήκατε από τους εθέρες και πήρατε το τρένο. Το δεύτερο θέμα σας σήμερα το βράδυ. Συχνά βέβαια οι πολιτικοί λένε ωραία λόγια, αλλά οι πράξεις υπολείπονται. Τα ίδια βλέπουμε και εδώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχουμε πολλούς και ωραίους στόχους. Ορισμούς τους επιτύχαμε, άλλους καθόλου. Ειδικά σε ό,τι αφορά την ενιαία αγορά και κυρίω των μεταφορών και κυρίω των σιδηροδρόμων, πολλά δεν έχουν επιτευχθεί ακόμα. Είχαμε καλέ προθέσεις και ίσω η Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση αυτή να αποδεικνύεται χάρτινο τίγρη ή δεν έχουμε την ικανότητα να πλασάρουμε το προϊόν. Αυτό που θέλουμε δηλαδή να περάσουμε στον κόσμο. Θέλουμε ανεξαρτησία, θέλουμε μια ρυθμιστική αρχή. Στη Γερμανία ομολογώ ότι οι σιδηρόδρομοι καλά τα πάνε. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν φτάσει στην καλύτερη δυνατή χρήση τους. Χρειαζόμαστε μια ρυθμιστική αρχή η οποία να μπορεί να κατανέμει τις διάφορες διαδρομές. Είναι τροπή βέβαια ότι από τις 27 χώρες μέλη, δύο, η Μάλτα και η Κύπρος που δεν έχουν καθόλου σιδηροδρόμους δεν έχουν και τίποτα να ε, μεταφέρουν στην εθνική του νομοθεσία. Αλλά άλλε χώρε όπω το Ηνωμένο Βασίλειο, όπω η Φιλανδία και ε, η Σουηδία έκαναν το καθήκον του. Μετέφεραν στην εθνική νομοθεσία. Όλε οι υπόλοιπε υπολείπονται. Και γι' αυτό βρίσκω ότι είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προβλέψει και μηχανισμού επιβολή κυρώσεων. Αλλιώ δεν πρόκειται ποτέ να μα πάρουν στα σοβαρά. Πρέπει να αντιληφθούν οι χώρε μέλη ότι όλε και όλοι θα υποφεληθούν από το άνοιγμα τη ε, Αγορά των σιδηροδρόμων. Όλοι βέβαια το λένε αυτό, όλοι τα λένε στα λόγια, δεν κάνουν όμως τα απαραίτητα έργα. Πρέπει να προχωρήσουμε λοιπόν και στα οικονομικά. Πρόσφατα στη Σαραγώσα διαπιστώσαμε ότι λείπουν οι πόροι, δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Πρέπει να απευθυνθούμε βέβαια στις χώρες μέλη να κάνουν κάτι παραπάνω. Ξέρουμε ότι για την ώρα με στην κρίση είναι δύσκολο αυτό, αλλά το χρειάζεται η Ευρώπη. Σας ευχαριστώ κυρία μου. Ακολουθεί εξ ονόματος των Πράσινων ο κύριος Κράμερ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το πρώτο πακέτο των σιδηροδρόμων κανονικά έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Μάρτιο του 2003. 22 χώρες μέλη ως τώρα δεν το έχουν εφαρμόσει. Μόλις τον Ιούνιο του 2008 ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γι' αυτό και πρέπει να την επιπλήξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίω και τι 22 χώρε μέν. Αλλά όπω λέω και την Επιτροπή που είναι θέμα των συνθήκων. Είναι απαραίτητη βέβαια να υπάρξει ανεξαρτησία των ρυθμιστικών αρχών. Οι τιμέ των ε, οι τιμολογίων πρέπει να είναι ξεκάθαρες. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, στο Βερολίνο, οι τιμές που πληρώνει ε, ο σιδηρόδρομος είναι διπλές από αυτές του Αμβούργου. Αυτά και αδιαφανή είναι και αυθαίρετα είναι και αντικονομικά εν τέλει. Είναι απαραίτητο να ανοίξουν τα δίκτυα. Είναι απαραίτητο επίση να ισχύσει αμοιβαιότητα. Δεν είναι δυνατόν ορισμένε χώρε να προστατεύουν του ιδιοδρόμους του και να προσπαθούν να μπουν στι αγορέ άλλων χωρών. Και εδώ λοιπόν απαιτείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω θεματοφύλακα των συνθηκών να επιβάλλει την τήρηση του υφιστάμενου δικαίου πρέπει να σταματήσει και ο αθέμητος ανταγωνισμός με τους άλλους τρόπους μεταφορών. Όταν στο σιδηρόδρομο επιβάλλονται διόδια σε κάθε μηχανή έλξης ανά χιλιόμετρο που διανύει, ενώ στους αυτοκινητοδρόμους είναι υπόθεση της κάθε χώρας να αποφασίσει αν θα επιβάλλει διόδια ή όχι. Αυτά τα πράγματα βεβαίως οδηγούν σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Από την άλλη μεριά, οι οδικές μεταφορές επιβαρύνουν πολύ περισσότερο το περιβάλλον και, τον και την ατμόσφαιρα από ό,τι ο σιδηρόδρομος. Παραπάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ δίνονται στην, ε, στις οδικές μεταφορές και στις ε, εναέρειες μεταφορές. Ενώ πολύ λιγότερο για την ε, επιδότηση των καυσίμων των σιδηροδρόμων. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν 85% των πιστοποιητικών εκπομπών καυσαερίων δωρεάν, ενώ ο σιδηρόδρομος αναγκάζεται να το πληρώσει. Χρειαζόμαστε λοιπόν θεμητό ανταγωνισμό, έντιμο ανταγωνισμό, όχι μόνο μεταξύ των σιδηροδρόμων, αλλά και μεταξύ των τρόπων μεταφοράς. Η Κομισιόν, που επαναλαμβάνει είναι θεματοφύλακα των σχετικών έχει πολλή δουλειά να κάνει και ας αρχίσει να το κάνει. Αν το κάνει, θα έχει σίγουρη την υποστήριξη του Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Κύριε Κράμερ, ο κύριος Ένα της ε, Ενωτικής Αριστεράς. Για τρία λεπτά. Η ελευθερία της μετακίνησης είναι από τα δικαιώματα των πολιτών και είναι απαραίτητο να μπορεί ο καθένας να έχει επομένως πρόσβαση σε ασφαλείς μεταφορές ποιοτικές και οικολογικές και οικονομικά προσιτές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει δίκτυο που εξυπηρετεί ολόκληρη την επικράτεια με καλές διασυνδέσεις. Άρα και πολύ καλούς σιδηροδρόμους δημοσίας ιδιοκτησίας ώστε να μπορέσει να καλύπτεται όλο η επικράτεια και να διασφαλίζεται η ποιότητα οι επιβάτες είναι πολίτες που έχουν δικαιώματα και δεν είναι απλώς πελάτες για τους οποίους μετράει μόνο το πάχος του πορτοφολίου. Το κοινοβούλιο μας δυστυχώς επέλεξε δογματικά τις σιδηροδρομικές μεταφορές να μην τις κάνει τα στήσει εργαλείο απελευθέρωσης αλλά μόνο ένα μέσο για οικονομική εκμετάλλευση. Έχουν καταστραφεί δίκτυα και υποδομές και έχει μειωθεί η ασφάλεια, έχουν απαγορευτεί οι επιχορηγήσεις, οι διασταυρωνόμενες επιχορηγήσεις που επέτρεπαν την κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας, ενώ παράλληλα δαπανήθηκαν εκατομμύρια για ατμομηχανές που μπορούσαν να που δεν είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν ολόκληρο το δίκτυο. Έτσι αυξάνεται η τιμή, κλείνουν οι γραμμές και καταστρέφονται οι υποδομές και κυρίως μειώνεται το επίπεδο ασφαλείας. Όταν διαχωρίσει κανείς τις ε, υποδομές από την υπηρεσία και θεωρήσει την ασφάλεια σαν ε, όχι πρωτεύον θέμα, ειδού που καταλήγουμε. Έχουν πολλαπλασιαστεί τα ατυχήματα και αυτή είναι μία από τις τρομερές αλλά επιπτώσεις της ανεύθυνης πολιτικής σας. Με την σιδηροδρομική δέσμη αντί να εξυγχρονιστούν οι ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι και να έχουν τα μέσα να ανταποκριθούν στους στόχους τους, γίνονται δευτερεύον τρόπος μεταφοράς και αυτό είναι ανόητο και άδικο και βλάπτει την εξυπηρέτηση των πολιτών με τη δέσμη αυτή γίνεται βραδύτερη συγκοινωνία από ό,τι πριν από 100 χρόνια. Μας λέγατε ότι ο ανταγωνισμός θα μειώσει τις τιμές, το αντίθετο έγινε. Όπως και για την ενέργεια ο ανταγωνισμός αύξησε τις τιμές για τον καταναλωτή και την καταναλώτρια. Και τελευταίο παράδειγμα, η γαλλική σιδηρόδρομοι που είναι κυρίως ηλεκτρικοί αγόραζαν με ειδική ταρίφα από τη δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού αλλά το 2011 προβλέπεται να πληρώνει 11% πιο ακριβά τον ηλεκτρισμό της. Ευχαριστούμε κυρία Επιτροπή και κύριε Ανταγωνισμέ. Ιδού τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ακολουθούν οι υπόλοιποι γεγραμμένοι συνάδελφοι για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι περιμένουμε αυτή την αναθεώρηση της δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμων εδώ και 20 χρόνια. Και αυτό αποτελεί σαφώς κακό παράδειγμα. Εχθές το Κοινοβούλιο ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο για μεταφορά επιρρουμάτων με στόχο να βελτιωθεί η κυκλοφορία στις βασικές, στους βασικούς ευρωπαϊκούς άξονες. Αυτό θα πρέπει να το διασφαλίσουμε μέσω ε, της άρσης όλων των φραγμών και των φυσικών αλλά και των διοικητικών φραγμών. Η αγορά θα πρέπει να γίνει ελεύθερη να μην υπάρχουν φραγμοί, να απλουστευτούν οι διαδικασίες και να υπάρχει μια πραγματική αγορά στην οποία θα υπερισχύει αμοιβαιότητα. Ο όρος αυτός χρησιμοποιήθηκε σε πάρα πολλές παρεμβάσεις ε, που ακούστηκαν πριν από μένα. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι ο διαχωρισμός ε, των υποδομών από τη διαχείριση είναι ένα θετικό βήμα. Είμαι πεπισμένος ότι οι επενδύσεις μέσω του, ε, των επενδύσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα είναι θετικό βήμα και όλα αυτά θα μπορέσουν να οδηγήσουν στη διαφάνεια, στην ελεύθερη αγορά και θα επιτρέψουν σε όλους να έχουν πρόσβαση σε μια αγορά η οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά έχει τεράστιες ανάγκες. Ειδικά αυτή τη στιγμή που διανύουμε μια περίοδο οικονομικών αναγκών και μέσω επενδύσεων καλά θα κάνει η Ευρώπη να ξεκινήσει και κάποια χρηματοδότηση ακριβώς ε, για να ε, παρακινήσει τον ιδιωτικό τομέα να επενδύσει και να ε, ανακτήσει το χαμένο χρόνο. Όλα αυτά βέβαια με ε, προστασία για το περιβάλλον και ασφάλεια και προστασία για τον ε, επιβάτη. Αυτά αποτελούν ε, αναπόσπαστο κομμάτι της όλης διαδικασίας, αλλά θεωρώ ότι ήγηκε και η ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει σαφώς στις ερωτήσεις μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπράιαν Σίμψον. Δύο λεπτά εκ μέρους των σοσιαλιστών. Κύριε Πρόεδρε, θα θυμάστε ότι σε προηγούμενες συζητήσεις εδώ στην αίθουσα που ε, είχα μιλήσει εκ μέρους της Επιτροπής Μεταφορών σας επεσήμενα πόσο ε, κακά είναι τα στατιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των σιδηροδρομικών μέτρων. Αυτό δείχνει και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα και στα κράτη-μέλη ότι όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει να εφαρμοστούν τα όσα συμφωνήσαμε, αλλά θα πρέπει να διασφαλίσουμε και ότι θα συμβεί αυτό. Το πρώτο πακέτο θα έπρεπε να είχε μεταφερθεί, όπως είπε και ο κύριος Φινάντς, από τα κράτη-μέλη το Μάρτιο του 2003. Το γεγονός ότι 22 κράτη-μέλη έχουν αποτύχει σημαίνει ότι ήταν πλημελή η προσπάθεια από πλευρά κρατών μελών και ανεξάρτητα από αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν και πάρα πολύ μικρή προσπάθεια εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Αυτό μα υπενθυμίζει πόσο πολλά εμπόδια παραμένουν όταν προσπαθούμε να εφαρμόσουμε μέτρα για του σιδηροδρόμους και αυτά θα πρέπει ε, να ισχύουν και εντό και εκτό τη σιδηροδρομικής βιομηχανία. Είδαμε μία επιχείρηση σιδηροδρόμων να πιέζει για την έκθεση για τους σιδηροδρόμους. Βέβαια απέτυχαν τεράστιες προσπάθειές τους, αλλά σημαίνει ότι προσπαθούν και ότι υπάρχουν και άλλες ε, σιδηροδρομικές εταιρείες στα κράτη-μέλη που ενδιαφέρονται για τα προσωπικά τους συμφέροντα και όχι για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει πρόοδο στο θέμα αυτό ουσιαστικά Ανακόπτηκε την ικανότητα των σιδηροδρομικών εταιριών της Ευρώπης να ανταγωνιστούν ε, τις άλλες εταιρείες ε, με ποιήσεις όρης και ακριβώς μας καταδεικνύουν πόσο ε, κατεπίγουσα είναι η ανάγκη να λάβουμε μέτρα. Θα πρέπει να έχουμε μια μακροπρόθεσμη προοπτική για τους σιδηροδρόμους μας και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν όλοι οι εμπλικόμενοι φορείς δεσμευθούν προς αυτό το στόχο. Περιμένουμε να τηρήσουν τα κράτη-μέλη τις ε, συμφωνίε τους και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τους πιέσει να τις τηρήσουν. Περιμένουμε δράση. Σήμερα είναι τα γενέθλια του κυρίου Κράμερ και ελπίζω να μπορέσουμε να του παραδώσουμε αυτή τη δέσμη μέτρων ε, εντός ε, της... όσο θα είναι ακόμα ζωντανός. Ε, ευχαριστώ. Συγχαίρουμε και εμείς ε, τον κύριο Κράμερ για τα γενέθλιά του. Ο κύριος Τούσας. πουλήματος του δημόσιου λαϊκού πλούτου και παράδοσης του στα χέρια των μονοπωλίων. Η επιβράδυνση εφαρμογή της ιδιωτικοποίηση των σιδηροδρόμων και της ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης απελευθέρωσης στι περισσότερε χώρε της Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποτέλεσμα των εργατικών λαϊκών αγώνων αλλά και των οξυμένων ενδοϊμπεριαλιστικών αντιθέσεων για το ποιο από τα μονοπόλια θα πάρει μεγαλύτερο κομμάτι των σιδηροδρομικών μεταφορών. οι εξελίξει στι σιδηροδρομικέ μεταφορέ στο ηνωμένο βασίλειο στη γαλλία τη γερμανία την ελλάδα και σε άλλα κράτη μέλη τη ευρωπαϊκή ένωση επιβεβαιώνουν τι εκτιμήσει μα. οι ελληνικοί σιδηροδρόμοι περικόπτουν τα δρομολόγια του στο όνομα τη εξυγίανση και στα πλαίσια των δεσμεύσεων από το μνημόνιο τη κυβέρνηση του πασόκ με την ευρωπαϊκή ένωση την ευρωπαϊκή κεντρική τράπεζα το διεθνές νομισματικό ταμείο αφαιρώντας το δικαίωμα της μετακίνησης σε κατοίκου και της μεταφοράς προϊόντων σε πολλές περιοχές της ελλάδας υποβαθμίζοντα τις δυνατότητες ανάπτυξης της χώρας. η υπερχρέωση του οσέ προκλήθηκε από την αντιλαϊκή πολιτική τη ευρωπαϊκής ένωσης και των κυβερνήσεων του πασόκ και της νέας δημοκρατίας τον εκφυλισμό του δημόσιου χαρακτήρα του σιδηροδρόμου και την μετατροπή του σε παράδεισο ιδιωτικών εργολαβικών συμφερόντων χρυσόφορο τομέα για την αύξηση των κερδών των μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων που λαιλάτισαν τον οσε. σήμερα η κυβέρνηση του πασόκ ετοιμάζεται να ξεπουλήσει τα φιλέτα του οσε να παραχωρήσει τις εκτάσεις του στο θριάσιο και άλλες υποδομές στα λιμάνια της ελευσίνας του πειραιά της θεσσαλονίκης και να επιδοτήσει τις επιχειρήσεις για τις άγονες γραμμές, σιδηροδρομικές γραμμές, εφαρμόζοντας την πολιτική ιδιωτικοποιήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις δεσμεύσεις που έχει κάνει στα πλαίσια του Μνημονίου. Το μεγάλο κεφάλαιο αντιμετωπίζει την κρίση σαν μια νέα ευκαιρία για να εξασφαλίσει και αύξηση των κερδών του από την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και των φυσικών πόρων και το ξεπούλημα της λαϊκής δημόσιας περιουσίας. Το ξεπούλημα του οργανισμού σιδηροδρόμων ελλάδας περιλαμβάνει πακτολό κρατικών επιθετήσεων αύξηση των ε, ατυχημάτων και πακτολό επιδοτήσεων σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους μαζικές απολύσεις και σαρωτικές αλλαγές σε εργασιακά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα των εργαζομένων. οι μεταφορές το σύνολο των υποδομών όπως και άλλοι στρατηγικοί τομείς της οικονομίας πρέπει να είναι λαϊκή περιουσία και να λειτουργούν προ όφελο τη εργατική τάξη και των λαϊκών στρωμάτων. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ κύριε Τούσα. Ήταν η τελευταία παρέμβαση. Α, όχι, ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, το ψήφισμα ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προωθήσει ακόμη περισσότερο και με εντονότερο και εντατικότερο τρόπο το σχέδιο αυτό για τους υδροδρόμους. Η εφαρμογή της υφιστάμενης οδηγίας δεν προσκόπτει μόνο στην έλλειψη θέλησης των χωρών μελών, αλλά και σε ορισμένες ασάφειες που εμπεριέχει. Ορισμένες χώρες μέλη βρήκαν εθνικές λύσεις, οι οποίες δεν παρεμποδίζουν ωστόσο την εφαρμογή της οδηγίας. Η πραγματικότητα και κυρίως η έλλειψη τεχνικής εναρμόνισης μεταξύ των χωρών μελών αλλά και τα διαφορετικά συστήματα ασφάλειας του τροχαίου υλικού δυσχεραίνουν την απρόσκοπτη διαμεθοριακή διακίνηση των σύρμων. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η κοινωνική διάσταση. Εδώ πρέπει να τεθεί το θέμα των συνθήκων εργασίας και των ελέγχων ασφαλείας. Επίσης το άλλο θέμα είναι τα σημεία εχμής στα σύνορα, στις μεθορίους, τα λεγόμενα bottlenecks. Εκεί πρέπει να ενισχυθεί η προσπάθεια για το, να ξεπεραστούν. Για παράδειγμα, μεταξύ Γερμανίας και Λουξεμβούργου. Εδώ και χρόνια συζητείται η διεύρυνση ε, ε, των υποδομών, αλλά εξακολουθούν λόγω των προβλημάτων να μην γίνονται οι απαραίτητε προσπάθειε. Εγώ θα ζητήσω λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με, τον, με την ίδια ζέση που προωθεί τον ανταγωνισμό να προωθήσει και τα άλλα θέματα τη εναρμόνιση δηλαδή των τεχνικών υποδομών και των συνθήκων εργασία και ασφαλεία. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ερχόμαστε στο Catch Η κυρία Τικάου ζήτησε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η Ένωση χρειάζεται μία μέθοδο συνδυασμένων μεταφορών διευρωπαϊκός και η σιδηρόδρομη είναι κάτι το ιδιαίτερα σημαντικό. Ζητούμε από τα κράτη-μέλη να δώσουν περισσότερη σημασία στις συνδρομικές μεταφορές χορηγώντας χρηματικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για τον εξυγχρονισμό των υποδομών τους. Η απελευθέρωση του τομέα των μεταφορών αυτών έχει αρχίσει. Το άνοιγμα των αγορών όμως δεν πρέπει να γίνει με απώλεια της ποιότητας ταυτόχρονα, ούτε της ασφάλειας ή της άνεσης των επιβατών και επιβατριών. Μόνο έτσι, από αυτές τις, από αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει πιο θελκτικός ο σιδηρόδρομος. Θα ήθελαμε λοιπόν να ζητήσουμε από την Κομισιόν κατά την επόμενη αναθεώρηση της δέσμης αυτής να συμπεριλάβει και ορισμένες κοινωνικές ρήκτρες ώστε να υπάρξουν πανευρωπαϊκά πρότυπα και σε εθνικό επίπεδο η κοινωνική περίθαλψη να υπάρχει και για όλους τους εργαζόμενους του σιδηροδρόμους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε συνάδελφε. Ακολουθεί ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μιλούμε για την εφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης των σιδηροδρόμων. Είπαμε ότι η μεταφορά στα εθνικά δίκαια δεν έχει γίνει θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μάλλον το 2003. Ε, μέχρι τώρα 22 μέλη δεν την έχουν επιτελέσει. Μήπως πρέπει να εξεταστεί εάν οι κανόνες εφαρμογής των οδηγιών της πρώτης δέσμης δεν είναι κατάλληλοι. Δεν είναι δυνατόν 22 χώρες μέλη να μην έχουν μεταφέρει. Ε, θα χρειαστεί ένας διάλογος μεταξύ της Επιτροπής και των Υπουργείων. Βεβαίω είναι ο κοινά επιθυμητό ο στόχος της βελτίωσης. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Θα δώσω τον λόγο πάλι στην Επίτροπο κυρία Γεωργίευα για να απαντήσει τις διάφορες παρεμβάσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. να ευχαριστήσω εκ νέου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πολύ χρήσιμη και συγκινησιακή συζήτηση που γίνεται επί του θέματος από καιρού καιρών. Διότι πράγματι όλοι θέλουμε όσο θα είμαστε εν ζωή να έχουμε ένα ε, καλός λειτουργών σιδηροδρομικό σύστημα και ελπίζω να ζήσουμε και αρκετά για να το δούμε. Στο παρελθόν συμμετείχα στην αναδιάρθρωση των σιδηροδρόμων δύο χωρών που πλέον ε, ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και γνωρίζω πράγματι πόσο δύσκολο είναι να προχωρήσει ένα σύστημα το οποίο έχει μακρά παράδοση κάποιες φορές, έχει σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό, έχει αντικρουόμενα συμφέροντα. Και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει όλοι να εμείνουμε στο ε, θέμα αυτό, διότι ένα ολοκληρωμένο και πολύ αποτελεσματικό σύστημα σιδηροδρόμων είναι απαραίτητο για την ευημερία των Ευρωπαίων, αλλά και για την ανταγωνιστικότητα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη τα σχόλιά σας και θα συνεχίσουμε να προωθούμε τις πρωτοβουλίες τις οποίες θέλουμε να πετύχουμε στον τομέα αυτό. Δεν είναι χάρτινος ο τίγρης. Αν κρίνουμε από τις διαδικασίες επιπαραβάση που έχουμε, γιατί καθυστέρησε τόσο η διαδικασία. Καθυστέρησε διότι υπήρχε μια διαδικασία ε, συζήτησης με τα κράτη-μέλη, υπήρχε και η διεύρυνση η οποία έφερε και νέα στοιχεία στο σύστημα και υπήρξε και μια απόπειρα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει κάποιο νόημα αυτή η συζήτηση με τα κράτη-μέλη, να αποστείλουμε συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, να αναλύσουμε τι απαντήσει πολύ προσεκτικά και από εκεί και πέρα να συνεχίσουμε σε μια διαδικασία παρακολούθηση με τα κράτη-μέλη, ώστε ε, το αποτέλεσμα ε, να έχει ε, κάποια βαρύτητα. Οι διαδικασίε επί δεν είναι στόχο και αυτό σκοπό. Θέλουμε να έχουμε ένα καλό σύστημα σιδηροδρόμων που θα μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερες, ε, πιο ασφαλείς ε, υπηρεσίες προς τους πολίτες μας που θα προσανατολίζονται στους καταναλωτές. Και ε, η αναθεώρηση του πρώτης δέσμης μέτρων για τους σιδηροδρόμους θα σχεδιαστεί κατά τρόπον ώστε να διευκολύνουμε την εφαρμογή των μέτρων αλλά και τον εξυγχρονισμό των σιδηροδρόμων. Θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις ως απάντηση σε σχόλια και ερωτήσεις που μου ετέθησαν. Η πρώτη αφορά στο επίπεδο ασφαλείας. Ο λόγος είναι κατηγορηματικός, ο νόμος είναι κατηγορηματικός και λέμε ότι το επίπεδο ασφαλείας έχει αυξηθεί από τότε που άνοιξε η αγορά. Αλλά επειδή μιλάμε για ζωές ανθρώπων εδώ, ένα ατύχημα και μόνο είναι παραπάνω από όσα θα πρέπει να έχουμε. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε αυτό το επίπεδο ασφαλείας. Επιπλέον, άκουσα δύο σχόλια που αφορούσαν την εφαρμογή των υποχρεώσεων ε, των δημοσίων υπηρεσιών. Θα ήθελα να τονίσω ότι η πρώτη δέσμη μέτρων δεν αποτελεί εμπόδιο σε κάτι τέτοιο. Αυτά όλα εφαρμόζονται σε ξεχωριστή νομοθεσία και επομένω υπάρχει δυνατότητα να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Θα ήθελα να μοιραστώ με το Κοινοβούλιο τους τρεις βασικούς στόχους μας και να σας πω κάποια πράγματα που έχουν ήδη υλοποιηθεί. Καταρχάς θέλουμε να ε, βελτιώσουμε την πρόσβαση στην αγορά και να είναι οι προϋποθέσεις πρόσβασης ε, πιο διαφανείς και χωρίς διακρίσεις. Δεύτερον, να βοηθήσουμε να υπάρξουν επενδύσεις και από το ε, δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα. Και τρίτον, κάτι το οποίο αναφέρεται πολύ από εσά, να ενισχύσουμε την ε, ρυθμιστική επιτήρηση των σιδηροδρομικών αγορών ώστε να έχουμε αγαστή συνεργασία μεταξύ των φορέων και να έχουμε και καλύτερες υπηρεσίες για όσους χρησιμοποιούν την υπηρεσία. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δεσμεύσει τους Υπουργούς να ξεκινήσουν ένα διάλογο επί του θέματος. Ε, οι Υπουργοί Μεταφορών έχουν εστιάσει την προσοχή του στου σιδηροδρόμου και θα φροντίσουμε να παραμείνει η προσοχή του εκεί και να βρίσκεται στη μερίσια διάταξη των θεμάτων που συζητούν. Σύντομα θα υιοθετήσουμε και την πρόταση αναδιατύπωση. Κατά πάσα πιθανότητα μέχρι το Σεπτέμβριο μπορεί να έχει παρουσιαστεί και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και προσβλέπουμε σε καλή συνεργασία μαζί σας για την μελλοντική νομοθετική διαδικασία και σαφώς να έχουμε απτά αποτελέσματα όσο θα είμαστε εν ζωή ή ακόμα νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ κυρία Επίτροπε. Μένουν πολλά να κάνουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.